για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Θα δώσουμε το λόγο στον ε, εισηγητή, θα δώσουμε μετά το λόγο ή στον ε, κύριο Άρια Κανιέτζε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Με πονάει μέση μου και δεν μπορώ να έρθω εδώ με την ταχύτητα που θα ήθελα. Πάλι συγγνώμη. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Τόρβελτς. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη για το έργο των συναδέλφων των σκιωδών εισηγητών. Υπήρχε πολύ ενδιαφέρουσα δυναμική στην ομάδα με συμμετοχή διαφόρων κομμάτων από διάφορες χώρες, διαφορετικές απόψεις, με διαφορετικές προτεραιότητες. Παρόλες τις διαφορές όμως δεθήκαμε στη διαδικασία. Και έχουμε γίνει και αρκετά καλοί φίλοι παρά τις διαφορές μας. Ακόμα και δεν είναι παρούσα προεδρία αυτή τη στιγμή, θέλω να ευχαριστήσω και την Προεδρία για τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε, διότι χωρίς την σημαντική συνεισφορά της, δεν θα τα καταφέρναμε. Ξέρω ότι το ξεκίνημα ήταν πολύ άσχημο στο Συμβούλιο. Έκαναν ό,τι μπορούσαν όμως. Και μετά από ψαξίματα καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο είναι, περιέχει πολλές τεχνικές λεπτομέρειες και πολλές ιδέες. Δύο πράγματα με ανησυχούν όμως. Θέλαμε να μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος. Δεύτερος, η Ευρώπη να ανοίξει για τεχνολογική πρόοδο. Δεν είναι πλέον ανοιχτή. Μετά τις ψηφοφορίες στην ΕΜΒΗ πρέπει να διερωτηθούμε. Πετύχαμε το στόχο μας. Η ειλικρινής απάντηση είναι όχι. Είχαμε πολύ υψηλότερους στόχους. Θέλαμε να μειώσουμε τα έργα του θερμοκηπίου. Η Ευρώπη να πετύχει τους στόχους του 2020, του 2030 και του 2050 ακόμα. Και ανησυχώ πάρα πολύ και νομίζω ότι και οι συνάδελφοί μου, οι σκιώδεις εισηγητές, αισθάνονται παρομοίως. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν πετύχαμε τους στόχους. Θέλαμε να ανοίξει η Ευρώπη όσον αφορά τη τεχνολογική πρόοδο. Σημαντικότατος ο στόχος αυτός κατά την απόψή μας, διότι αν δεν προχωρήσει τεχνολογικά η Ευρώπη, η Ευρώπη θα μείνει πίσω θα υποβαθμιστεί σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη θέση στον κόσμο όσον αφορά αυτά τα θέματα. Έχουμε συστημικά λατώματα, έχουμε ε, μια αναστέλουσα μειοψηφία στο Συμβούλιο και καμιά φορά αυτή διαμορφώνεται στη δικτατορία της μειοψηφίας. Έχουμε κράτη-μέλη που φοβούνται το μέλλον. Και όταν φοβούνται το μέλλον τα κράτη-μέλη δεν τολμούν να λάβουν τις σωστές αποφάσεις σηκώνουν το χειρόφρενο και προσπαθούν να κινηθεί η Ευρώπη με το χειρόφρενο. Αυτά είναι τα προβλήματα όσον αφορά τις εργασίες του Συμβουλίου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε. Αν το Συμβούλιο δεν μπορεί να δει τι θα γίνει στο μέλλον, αν το Συμβούλιο δεν μπορεί να δει το φως στον ορίζοντα, τότε δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας αλλά θα δευτερολογήσω αφού ακούσω τις απόψεις των ε, σκιωδών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα έχει τον λόγο ο κύριος Αρίας Κανιέντε. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί κύριοι βουλευτές, για μένα είναι πάρα πολύ ευχάριστο να συζητάμε τώρα. Ε, να συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση για τα κάψιμα και τώρα βρισκόμαστε ενώπιον μια συμφωνία Οπότε έτσι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το, αυτό το υλικό και να υποστήριξουμε και τη βιομηχανία. Για μα είναι ξεκάθαρη αυτή η πορεία όσον αφορά αυτού του είδου τα βιοκαύσιμα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και επίση γνωρίζω ότι αυτή η πορεία δεν ήταν εύκολη. Οπότε γι' αυτό και είμαστε υπέρ αυτή τη συμφωνία να ολοκληρώσουμε τι διαπραγματεύσει και θα πρέπει βέβαια να ευχαριστήσουμε όλους τους βουλευτές, ακόμη και εκείνους οι οποίοι και στην προηγούμενη θητεία ε, δούλεψαν τόσο σκληρά για αυτή την υπόθεση. Επίσης πρέπει να ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Τόρβαλτ και τον κύριο Λαβία και την ομάδα διαπραγματεύση γιατί κατέβαλαν προσπάθειε ούτω ώστε να φτάσουμε στην τελική ευθεία. Αυτός ο συμβασμός είναι ε, προϊόν κάποιων υποχωρήσεων και γιατί υπήρξε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε πολλές ε, ευκαιρίες ώστε να βρούμε τα σημεία συμφωνίας. Αυτή η δέσμη διατάξεων που έχουμε είναι πάρα πολύ αξιόλογη. Το... Και η πρώτη ανάγνωση επίσης πήγε καλά όσον αφορά ε, <clears throat> το Κοινοβούλιο. Και τώρα έχουμε εδώ πέρα τα βιοκαύσιμα από κάποιες καλλιέργειες. Και αυτό θα γίνει με ρύθμιση της ε, οδηγίας για τις χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εμείς ε, καταρχήν είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, μια οροφή 5% δηλαδή το μισό του στόχου που έχουμε για την ανανεώσιμη ενέργεια στον αφορά τις μεταφορές. Και αυτό το επιλέξαμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις πηγές, τις συνεργέ που έχουμε τώρα και να υποστηρίξουμε την ε, βιομηχανία. Οπότε τελικά ε, το 5% έγινε 7%. Ανέβηκε παραπάνω σαν συμβασμός και αυτό είναι παραπάνω από όσο στην αρχή προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως αυτό μπορεί να ε, ρυθμίσει το πόσο θα χρησιμοποιηθεί το iLook. Τώρα, με αυτόν τον συμβασμό θέλουμε να πετύχουμε την μετάβαση σε βιοκαύσιμα πιο προοδευμένα. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει για τα βιοκαύσιμα να ορίσουν ένα στόχο του επίπεδου του 0,5%. Αυτό δεν είναι δεσμευτικό, αλλά έχουν κάποιο προορισμό τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να ορίσουν αυτό το επίπεδο στο οποίο θέλουν να φτάσουν για τα ε, πιο προθυμένα βιοκαύσιμα. Και έτσι θα πρέπει να έχουμε μια ρεαλιστική λύση. Και ελπίζω ότι πέραν το, του ορίζοντα 2020 και τα άλλα πράγματα που έχουμε, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Επίσης, με αυτούς τους συμβασμούς τώρα θα έχουμε βελτίωση όσον αφορά την καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Και θα έχουμε τώρα κάποιες ε, εγκαταστάσεις που θα δουλεύουν με 60% εξοικονόμηση ενέργεια σε σχέση με τα παραδοσιακά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το iLook έχει υπολογίσει κάποιες τιμές οπότε θα έχουμε κάποια έκθεση η οποία θα, θα μας δώσει το τι βλαπτικά αέρια θα παραχθούν και ε, είχαμε έρθει σε ε, αντίθεση με τη θέση του Συμβουλίου, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με εφορμή την οδηγία για την ενέργεια από πηγές. Πάντως τώρα, εκεί που καταλήξαμε, ήταν ένα βήμα πρόοδο. Και έτσι τώρα, αυτή η δέσμη των μέτρων θα μας επιτρέψει στη χρήση του άλλου και θα έχουμε αυτά τα προχωρημένα βιοκαύσιμα. Οπότε έτσι θα μπορούμε να ανατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Όλα όσα είχατε πει στην πρώτη ανάγνωση αντικατοπτρίζονται σε αυτό το τελικό κείμενο. Υπήρξαν δυσκολίες γιατί ήταν περίπλοκο το θέμα, αλλά νομίζω ότι αυτά τα οποία πέτυχε το Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστούμε κύριε πίτροπε Και τώρα έχουμε τις ε, παρεμβάσεις των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Πρώτα-πρώτα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να τράξω την ευκαιρία και να ευχαριστήσω τον κύριο Τορβάλτσα για το εξαιρετικό έργο που έκανε στην εκθέση αυτή. Εγώ ήμουν ε, πριν από 11 χρόνια καινούργιος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τότε διαπίστωσα ότι ο στόχος για τις ανανεώσιμε ήταν πάρα πολύ χαμηλός και ότι η πρόοδος ήταν πάρα πολύ αργή για την προώθηση των στόχων αυτών. Τώρα πλέον, στη Σουηδία, οι σοσιαλδημοκράτες, το κόμμα για το περιβάλλον, μιλάμε για εθανόλη, German, though. Sorry for... Μία διακοπή. Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω γερμανικά, όχι αυτή την ώρα το πρωί, δεν πάση περιπτώσει. Να το ξαναπροσπαθήσω. Είναι διαφορετική λοιπόν η κατάσταση σήμερα. Μιλήσαμε για την εθανόλη, τότε λες και ήταν ο δρόμος προς την κόλαση. Κοιτώντας ε, τους πράσινους, τους σοσιαλδημοκράτες, εδώ μιλάμε για τους στόχους μέσα από τις ανανεώσιμες. Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν αντλίες πετρελαίου που κάθονται και σκουριάζουν. Δεν μιλάμε όμως για το σενάριο της εθανόλης. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τα καύσιμα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε ένα πιο ευνοϊκό σενάριο. Η... Τα βιοκαύσιμα είναι σημαντικό συστατικό σε χώρες όπως η Σουηδία, για παράδειγμα, όπου χρειάζεται και χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα. Υπάρχει φυσικά κίνδυνος να πάει να τα πράγματα στραβά με την νομοθετική αυτή πρόταση και πολλές αξιώσεις ε, τίθενται, ιδιαίτερα από τους πράσινους και τους αριστερούς, γιατί μιλάμε για όρια σε ό,τι αφορά τη χρήση ε, των βιοκαυσίμων και Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε κανόνες και όσοι διατείνονται ότι είναι πράσινοι θα πρέπει να υπερψηφίσουν αυτή τη νέα πρόταση γιατί ιδάλλως υποστηρίζουμε τα ρεκτά καύσιμα. Ο κύριος Ντάνς, ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Τόρβα στον συγκεκριτή για τη δουλειά που έκανε. Πολύ συχνά ήταν δύσκολε οι περιστάσει που επικρατούσαν. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε να φτάσουμε εδώ, να πετύχουμε συμβιβασμό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που έκανε. Νομίζω ότι είναι σημαντικότατο έτσι μια στιγμή να δούμε γιατί διεξάγεται τη συζήτηση αυτή και γιατί το θέμα ήταν τέτοιο και αμφισβητήσιμο. Επί σειρά ετών βλέπετε, βλέπουμε τα αποτελέσματα κακής πολιτικής, ιδιαίτερα κακής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα βιοκαύσιμα. Αυτές οι συνέπειε είναι καψίδα και εγώ μόνος μου δουλεύοντας σε ΜΚΟ προηγουμένως, σε τομείς κυρίως σε περιοχές όπως είναι η Ποσαχάρια Αφρική, όπου κοινότητες υπέφεραν από πολύ ασχήμα αποτελέσματα των πολιτικών που εθετούσαμε εδώ κυρίως για τη διάδοση των ε, προϊόντων, για των καλλιεργιών, για παραγωγή βιοκαυσίμων εδώ, αντί να, παράγονται, να παράγονται τρόφιμα εκεί. Η ζωή των τοπικών κοινοτήτων εξαρτώταν από, αυτές, από αυτά τα εδάφη και οπότε και άλλαξε η χρήση της γης, άλλαξε το οικοσύστημα γιατί αλλάξαμε τις καλλιέργειες και αν δεν είχαμε κάνει αυτή την αλλαγή ε, ίσως να μην είχαμε τα προβλήματα της αλλαγής του, της ζωής εκεί. Λοιπόν, έχουμε ένα πακέτο μπροστά μας, έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις, θα το κρύψω, κυρίως για το στόχο για τα βιοκάψιμα πρώτης γενιάς που ε, θέλαμε τα επίπεδα να είναι πολύ πιο χαμηλά και αυτό το πακέτο αντικα το τοπτίζει κυρίως την αμετάκλητη θέση, αμετακίνητη θέση κάποιων κρατών μελών. Και αυτό φαίνεται κυρίως στη θέση που θετήθηκε από το Συμβούλιο και ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτή η θέση. Υπήρξε έλλειψη φιλοδοξίας, αν επιτρέπεται να το πω αυτό, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. παρόλα αυτά, αυτό που έχουμε είναι ένα βήμα προόδου και πρέπει να δεχτούμε ότι είναι κάτι σημαντικό. Είχαμε αδιέξοδο επί μακρών και δεν ήταν επωφελές για τις κοινότητες που προανέφερα, για τους ανθρώπους, ούτε ήταν επωφελές για τις βιομηχανίες που έχουν τις βέλτιστες προθέσεις και έχουν κάνει επενδύσεις εδώ και πολλά χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση. Και στο πακέτο αυτό επιτέλους διαλέγουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει έμεση αλλαγή της χύσεως των γεών και δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια βάση ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει ε, τα επιστημονικά δεδομένα που εκείνοι που ήταν αντίθετοι μας εμπόζουν να τα χρησιμοποιήσουμε. Κάποιοι αρνούνται τα αρνητικά αποτέλεσματα το, της χρήσης των βιοκαυσίμων και άλλοι μπορεί να εκμεταλλεύονται τη συμφωνία για να πετύχουν πόντους. Νομίζω ότι η συμφωνία είναι μεν ατελής αλλά αποτελεί βέμα πρόοδου και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Sí. Eh, señor Dank, tiene una tarjeta azul del señor Glesos. ¿La acepta? Έχει σηκωθεί Κύριε έχετε λόγο, κύριε ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο εάν γνωρίζει ότι ο τελευταίος σεισμός που έγινε στα Ιμαλάια έχει σχέση με την κλιματική αλλαγή η οποία συνεπιφέρει η οποιαδήποτε επέμβαση του ανθρώπου στη φύση και ιδιαίτερα γύρω από τα καύσιμα. Πολλά είναι τα αίτια των σεισμών, πιστεύω. Και τα τεκτονικά θέματα μετακίνηση των πλακών ίσως είναι το βασικό αίτιο αλλά θα είμαι έτοιμος να ακούσω στοιχεία για το πώς μπορεί να συμβάλλει η πολιτική των βιοκαυσίμων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις καταστροφικές σεισμικές δονήσεις του Νεπάλ. Αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία θα ήθελα να τα ακούσω. Είμαι ανοιχτό εγώ. Α το θέσω έτσι. Είμαι ανοιχτό σε αυτή τη θεωρία. Σα ευχαριστούμε. Και μετά από αυτή τη, μικρή δόση επιστημίου φαντασία, δίνουμε τώρα το λόγο στην κυρία Γκέρλινγκ, η οποία όμως δεν βρίσκεται στην αίθουσα και δίνουμε το λόγο στον κύριο Γκέρ Μπράντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Τόρβαλτς, για την εξαιρετική του δουλειά. Σίγουρα το μονοπάτι που χαράσει εδώ στο Κοινοβούλιο και που υπήρχε ήδη και οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο την οποία ξεκίνησε και κληρονόμησε ο κ. Στορβάλτς από την συνάδελφα του Κορίν Λεπάζ, είναι κάτι το οποίο δεν μας υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Γιατί μιλάμε μόνο για τους στόχους του 2020, τους στόχους για το κλίμα, το 20%. Αν μπορούμε Να φανταστούμε ότι σε κάποια χρόνια θα πρέπει να κινηθούμε προς το 80% μείωση του διεξιδίου του άνθρακα. Είναι λοιπόν δύσκολο το μέλλον, προδιαγράφεται. Κάνουμε πολύ πολύ μικρά βήματα και ε, υπάρχει μεγάλος πόλεμος. Τι θα γίνει αν θα χρειαστεί να κάνουμε μεγάλα βήματα. Είμαι πεπισμένος ότι δεν θα προχωρήσει η κλιματική πολιτική και εμείς στην Ευρώπη περηφανευόμαστε ότι θα πετύχουμε τους στόχους το 2020 και κοιτώντας τι γίνεται στη χώρα μου, την Ολλανδία. Και βλέπω τώρα ότι η οικονομική ανάπτυξη κάπως ξεκινάει Και αυξάνονται λοιπόν αυτόματα οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε πολύ. Ένα άλλο θέμα. Αυτή η μικρή προσαρμογή των δύο οδηγιών για την ποιότητα των καυσίμων και τι ανανεώσιμε. Η καλή πολιτική απαιτεί τόλμη, ιδιαίτερα σήμερα. Και ιδιαίτερα αν ε, η σημερινή πολιτική ξεπεραστεί από την επιστήμη. Γιατί φαίνεται ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική μας και θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι τα βιοκαύσιμα δεν είναι το ιεροποτήρι το οποίο υποστηρίζαμε ότι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Θα πρέπει όμως να υπάρχουν και κριτήρια βιωσιμότητας, να μην κάνουμε τα ίδια λάθη όπως πριν από κάποια χρόνια. Αλλά, επαναλαμβάνω, θα υπερψηφίσω το αποτέλεσμα, αλλά είναι πραγματικά πολύ συχνό, Πρόεδρε. Η συνάδελφος Κονέτσνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κυρίε. και κύριοι, όταν μετά τον τριμερή διάλογο σκεφτόμουν πώς να ψηφίσω για το τελικό κείμενο, είχα ε, μια αίσθηση απέραντης θλίψης. Ε, όλοι το ξέρουμε σήμερα ότι τα βιοκαύσιμα και η υποστήριξή τους ήταν ένα πολύ προβληματικό ζήτημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα μεγάλο λάθος. Πολλά στοιχεία παραγνωρίσαμε τότε και αυτό ε, υποβάθμισε το τοπίο μας και δημιούργησε κρίση τροφίμων. Είχα μεγάλες προσδοκίες ως κοιόδης εισηγήτρια για το σχέδιο αυτό. Δυστυχώ δεν μπορώ να πω ότι εκπληρωθήκαν. Καταρχάς υπήρχε καθημερινή πίεση από το, τα ευρωπαϊκά λόμπι για το ποιο καύσιμα θα επιδοτούταν και το καθεξής παρά το γεγονός ότι και ο εισηγητής και η Επιτροπή ΕΝΒΗ κάναμε δουλειά. Μπήκαμε στις τελικές διαπραγματεύσεις με ένα ισχυρό κείμενο. Το, το κείμενο όμως τελικά που προέκυψε ήταν πραγματικά ένα αποτέλεσμα πάρα πάρα πολύ δυναμό. Ουσιαστικά υποκύψαμε στις πιέσεις του Συμβουλίου. Χάσαμε το όριο του 6% για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς. Δεν μπορέσαμε να έχουμε επαρκή υποστήριξη για δεύτερη γενιάς βιοκαύσιμα, επιτρέποντας μη δεσμευτικούς στόχους. Και τελικά το Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να περάσει σχεδόν τίποτα από αυτά που πέρασαν στην ΕΜΒΗ. Ουσιαστικά το τελικό κείμενο είναι μόνο ελαφρώς βελτιωμένο σε σχέση με την πρόταση του 2009, μετά από πέντε χρόνια δηλαδή διαπραγματεύσεων δεν πετύχαμε κάτι πολύ καλύτερο. Και έτσι η Γκουέντζιέλ δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή τη φάρσα που ουσιαστικά επιτρέπει να συνεχιστεί το status quo. Κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστεί η υποβάθμιση του τοπίου μας και οι εταιρείε θα συνεχίσουν να υποφελούνται και αυτό μόνο σε εμάς οφείλεται. Κύριο Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή τον κύριο Τόρβαλτς για τη δουλειά που έκανε. Όπως προαναφέρθηκε δεν ήταν εύκολο θέμα, κυρίως για να δημιουργηθεί πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και να προχωρήσει και διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο και ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε. Τούτων λεχθέντων είμαι απογοητευμένο για τα αποτελέσματα. σω να είμαι πιο απογοητευμένο διότι το Συμβούλιο δεν είναι καν παρόν στι συζητήσει. Και αυτό δείχνει λίγο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή, εντό του Συμβουλίου τα κράτη-μέλη δεν βλέπουν το πρόβλημα καν. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ κακό μήνυμα που στέλνουν, δηλαδή ότι δεν ενδιαφέρονται. Και αυτό το είδαμε και σε πραγματεύσεις, ήταν ξεκάθαρο ότι ε, δεν ενδιαφέρονται και είναι πρόβλημα αυτό. Διότι γιατί κουβεντιάζουμε το θέμα. Θέσαμε ένα στόχο στα 10% για τα βιοκάψιμα στη, στον τομέα των μεταφορών. Όλοι γνωρίζουμε όμως ότι αν δει κανείς το πώς εξελίσσεται η κατάσταση Κυρίως βλέπουμε ότι αναπτύσσονται τα αγροκαύσιμα, βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς, τα οποία δεν δίνουν τα ωφέλη για το κλίμα που υποτίθεται ότι έπρεπε να πετύχουν. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πρόταση, προσπαθήσει να βάλει στο 5% το όριο για την πρώτη γενιά. Στο Κοινοβούλιο καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία σε ένα όριο του 6%, αλλά και τα κράτη-μέλη ήθελαν να είναι 7%. Δυστυχώς τις διαπραγματεύσεις χάσαμε αυτή τη θέση και στο τέλος σαν κοινοβούλιο συμφωνήσαμε με το 7%. Κατά την άποψή μου αυτό πόρο απέχει, είναι πολύ ψηλό, διότι καλύπτει το στόχο με τα κακά βιοκαύσιμα που δεν είναι εκείνα που θέλαμε να προωθήσουμε, τα πιο προχωρημένα βιοκαύσιμα. Αυτό ήταν το δεύτερο αίτημα του Κοινοβουλίου. Θέλουμε προωθημένα βιοκαύσιμα, τόσο ώστε πραγματικά να έχουμε καινοτομία στην Ευρώπη. Δυστυχώς και εδώ το Συμβούλιο δεν ήθελε τίποτα από όλα αυτά και στο τέλος έχουμε μη δεσμευτικό στόχο για τα προχωρημένα αυτά βιοκαύσιμα. Άρα είναι πολύ αδύναμο το μήνυμα ε, για την τόνωση της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δείτε τους ε, ορισμούς, και εκεί οι ορισμοί είναι αόριστοι, αρκετά αόριστοι. Πιθανότατα θα γίνει συζήτηση και όλοι θα θεωρήσουν ότι αυτά είναι προθυμένα καύσιμα, βιοκαύσιμα. Και όλοι το χρησιμοποιούν σαν νέα μόδα αυτά τα προχωρημένα βιοκαύσιμα, δεν θέλουν την καινοτομία. Και η έμεση αλλαγή τη χρήση των γιών είναι άλλο πρόβλημα. Θέλουμε αυτό να ληφθεί υπόψη. Ποια είναι η έμεση αλλαγή τη χρήση γιών. Λοιπόν, και δεν υπάρχει πραγματικό έλεγχο. Έχουμε υποβολή αναφορών και έχει πραγματικό έλεγχο. Χάσαμε πολλά, χάσαμε πολλά σαν κοινοβούλιο και γι' αυτό δεν υποστηρίζω τη συμφωνία αλλά βλέπω τον Επίτροπο που είναι παρόν και τον ρωτώ τι θα κάνουμε μετά το 2020. Θα μάθουμε από το πρόβλημα ότι δεν καθορίζουμε ένα νέο στόχο που είναι εντελώς άκαμπτος, αλλά πραγματικά βάλουμε, βάζουμε στο επίκεντρο την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων και θέτουμε σαν ένα στόχο για την μείωση αυτού και δεν έχουμε τεχνολογική φύση στόχο, διότι δεν ξέρουμε πώς θα αναπτυχθεί η τεχνολογία. Οπότε το θέμα είναι, θα συνεχίσουμε μετά το 2020 με την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, διότι τότε θα διεξαχθεί νέα συζήτηση και ελπίζω τότε να είναι παρόν το Συμβούλιο. Ήταν σημαντικότατο θέμα. Και αν κινηθούμε σωστά, πραγματικά θα έχουμε μια μεγάλη εναρμόνιση στον τομέα των μεταφορών. Αν κάνουμε λάθο όμω, θα τονώσουμε λάθο τεχνολογίε και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Κύριε Αϊκάουτ, δύο μπλε κάρτε έχουν ζητηθεί από τον Αποδέχεστε? Ορίστε, έχετε το λόγο. Κύριε Σάντζη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κάλτ, θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Συμφωνώ 100% ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει. Όμως, θα πρέπει να συμφωνήσουμε για την πρώτη, τη δεύτερη ή οποιαδήποτε τέλος πάντων η οποιαδηποτε τέλο παντων η γενια των καυσίμων. και σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει με τα ορυκτά καύσιμα. Μπορείτε τώρα να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση και μετά στην άλλη. Αν ε, νομίζω θα απαντήσω και στις δύο ερωτήσεις. Πρώτα πρώτα, όσον αφορά τα βιοκαύσιμα, θέλω να σα πω ότι δεν είναι η μόνη εναλλακτική λύση τα εναλλακτικά καύσιμα. Και ακριβώ αυτό είναι το θέμα. Ότι τώρα ε, έχουμε κλείνει προ ε, αυτή την εναλλακτική λύση, τόσο στι μεταφορέ, να ακολουθήσουμε αυτή την πολιτική. Οπότε, το, εστιάζουμε προσοχή μα μόνο σε μια πολιτική. Αυτό είναι χαζό. Ε, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δούμε πώς θα πετύχουμε το να μην έχουμε ε, διοξίδιο του άνθρακα μεταφορές και κατόπιν να δούμε τις ανελεκτικές λύσεις. Να μην επικεντρωνόμαστε μόνο σε μια κακή τεχνολογία η οποία ε, δεν αποδίδει. Και οπότε τι, θα στραφούμε στα ορυκτά καύσιμα, όχι. Γιατί ακριβώ να προσέξουμε, μην στραφούμε σε κάποια εναλλακτική λύση ακόμα χειρότερη για το περιβάλλον. Οπότε αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Και δεν νομίζω ότι προς το παρόν κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Χέλνερ. ευχαριστώ πολύ. Είπατε ότι εστιαζόμαστε υπερβολικά στα βιοκαύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνείτε ότι οι πράσινοι φταίνε γι' αυτό και ότι αυτή το πρόθεσαν πριν από 10 χρόνια αυτό. Κατά δεύτερον, είπατε τα βιοκαύσιμα. Τα αγροτικά δεν, έχουν, δεν επιφέρουν τα αποτελέσματα. Ξέρετε ότι Παράγουμε εθανόλη με πιστοποίηση μείωση 90% διοξιδί του άνθρακα και ότι μιλάμε για διαφορετικά βιοκάψαμα και τρίτον ότι αν το Κοινοβούλιο καταψηφίσει την ε, νομοθεσία αυτή αν είχατε ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα τολμούσατε να την επενδύσετε στην παραγωγή προηγμένων δεύτερης γενιάς βιοκαυσίμων αν το Κοινοβούλιο αποφασίσει να σκοτώσει και τους κανόνες αλλά και τους ορισμούς για τη χρήση τους. Κατά πρώτον κύριε Φιέλνερ, εγώ υπερψηφίζω της εντολής ΕΝΒΗ. Ξέρω ότι ήσασταν κατά. Δεν θέλετε τίποτα. Θέλετε υψηλότερο κατόφλι για τις νέας γενιάς. Εσάς έχετε, σας έχετε πουληθεί στο λόμπι των, ε, εδώ και καιρό. Το ξέρουμε αυτά. Αν θέλατε κάποια αλλαγή, θα είχατε συμμετάσχει στην ε, συμφωνία της ΕΝΒΗ. Εσείς στην διαπραγματεύσεις σας με τα πουλήσετε όλα. Τώρα υποκρίνεστε ότι είστε στην πλευρά του καλού. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να έχετε ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς. Κατά δεύτερον, αν θέλετε να κάνετε διάκριση μεταξύ καλού και κακού, γι' αυτό θα πρέπει να λάβετε υπόψη ε, την αλλαγή χρήσης. Γιατί αν δεν ληφθεί υπόψη, δεν ξέρετε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Γι' αυτό λοιπόν ε, προτείνω να ληφθεί υπόψη το iLog. Εσείς δεν το θέλετε καν. Εσείς θέλετε ένα στόχο που θα προωθεί τη γεωργία και όχι το καλό. Αν ήμουν εγώ παραγωγός ε, βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συμφωνία και διακόπτει ο πρόεδρος, όχι, συνεχίζει ο κύριο Εκάουτ. Είπαμε μέχρι ένα λεπτό. Ε, ε, γιατί θα σα κόβω το μικρόφωνο αν το υπερβαίνετε. Τέλος πάντων, ο κύριος Πεντιτσίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή τον κύριο Ντόρβαλτ για τι προσπάθειε που κατέβαλε μέχρι τώρα. Δυστυχώ όμω αυτό ο συμφιβασμό δεν μα ικανοποιεί καθόλου. Αντίθετα μάλιστα κατά τα λοιπά θα πρέπει να είναι δύσκολο να θεωρηθεί σαν συμβιβασμό. Διότι ε, πραγματικά μάλλον είναι προσπάθεια επιβολή θέσεω του Συμβουλίου που δεν θα αναλάβει ούτε κατ' ελάχιστον υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου, άρα και τη θέση των Ευρωπαίων πολιτών. Εμείς πολεμήσαμε για να υπερασπιστούμε όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που είναι παράδειγμα της κυκλικής οικονομίας. Αλλά η κυκλική οικονομία δεν ενδιαφέρει πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώ για εκείνες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ε, το χάρη και τα, τα απορρίμματα των ξύλων, της ξυλίας για να φτιάξουν έπιπλα. Ε, με αυτή την οδηγία θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα απόβλητα για την, για την παραγωγή βιοκαυσίμων προθυμένων. Ε, έβλαψε ε, την πρόταση του Κοινοβουλίου το Συμβούλιο και αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν την πρώτη ύλη και θα υποστούν την, τον του ανταγωνισμό τη βιομηχανία των προθυμένων βιοκαυσίμων. Ξέρετε πόσε επιχειρήσει μιλάω, για πόσε μιλάω, πάρα πολλέ επιχειρήσει μιλάω. Μιλάω για επιχειρήσει που κλείνουν τώρα. Ξέρετε πόσοι άνεργοι παραπάνω θα υπάρξουν λόγω αυτού του ανταγωνισμού όσον αφορά την πρώτη ύλη. Λοιπόν, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να προχωρήσει γρήγορα για, προς την απανθράκωση, την ε, μείωση της ίσως του άνθρακου στον τομέα και η νομοθεσία των βιοκαυσίμων να γίνει πραγματικά βιώσιμη και πραγματικά πράσινη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Έχετε μια μπλε κάρτα. Από την κυρία Γκραπίνη. Αποδέχεστε. Μάλιστα. Έχετε το λόγο κυρία Γκραπίνη. Ε, Αγαπητέ συνάδελφοι. Είπατε ότι αν τελικά αυτή ε, η πρόταση εγκριθεί θα επιβληθεί ανταγωνισμός σε εκείνους που παράγουν ενέργεια από το ξύλο, από την ξυλία. Θεωρείτε ότι δεν χρειαζόμαστε τελικά ανταγωνισμό στις οικονομίες μας. Ο κ. Φεντατσίνη. Σίγουρα χρειαζόμαστε ανταγωνισμό, αλλά δεν χρειαζόμαστε ανταγωνισμό αθέμητο. Μιλάμε για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτά τα απόβλητα της πρώτης ύλης, άρα ανακυκλώνουν την οικονομία και πρέπει να τη στηρίξουμε. Είναι θέμα προτεραιότητα. Εάν βγάλουμε την πρώτη ύλη από τι επιχειρήσει που ήδη πεθαίνουν, διότι ήδη έχουν πρόβλημα λόγω τη κρίσεω, και του βγάλουμε και του πάρουμε την πρώτη ύλη, θα έχουμε επιδείνωση από πλευρά απασχόληση και επιδείνωση τη ποιότητα του είδου των επιχειρήσεων που κανονικά θα έπρεπε να υποστηρίζουμε. Chers collègues, nous aurions tort de renoncer brutalement aux agrocarburants de première génération. Ναι, σωστό είναι το να θέλουμε να καταλήψουμε εδώ τα βιώσιμο πρώτης ε, ε, πρώτη γενιά και τότε της, ε, πέρσι είπαμε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τη χρήση της γέας και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απότομα διάλεξε ε, να, να, ε, να τροποποιήσει τέλος πάντων αυτές οι ιδέες του 1998 και του, και Οπότε τώρα θα έχουμε αυτές τις ε, επενδύσεις και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους γεωργούς μας οι οποίοι θεώρησαν ότι έτσι μπορούν να κάνουν κάτι για την κρίση που τους έχει χτυπήσει. Οπότε τώρα έχουμε τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς αλλά που όμως από ό,τι φαίνεται ακόμα δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν την πρώτη γενιά αυτά. Έχουμε αυτό το όριο το οποίο πρότεινε το Συμβούλιο. Νομίζω ότι είναι λογικό επί τη βάση των επενδύσεων των μακροπροθέσμων που έχουν γίνει. Και, ε, έχουμε τον νόμο πάρτου του 1923 και από τότε η Γαλλία ε, είναι πρωτοπόρα στα δύο καύσιμα, οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε στο παράδειγμα προς ε, μίμηση, αλλά να μην δυναμητίζουμε τις προσπάθειε. Señor Lise. Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν για τη συμβιβασμό αυτό και ιδιαίτερα τον κύριο Τόρβαλτς, τον Κρίστοφερ Φιέλνερ. Πιστεύω ότι είναι καλός συμβιβασμό και το ΕΛΚ θα υποστηρίξει τον συμβιβασμό αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει μια μετακίνηση μετριοπαθής, αλλά να μην τα πετάξουμε και τα τενάξουμε όλα στον αέρα. Ούτε είναι καλό σήμα προς τους ε, αγρότες και προς όλους που όσοι επένδυσαν μετά από χρόνια να πούμε ότι α, όλα ήταν λάθος. Υπάρχει και προστασία της εμπιστοσύνης. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι η πολιτική των βιοκαυσίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αιτία όλων των προβλημάτων σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει υπερβολική ε, δραματοποίηση της κατάστασης. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να αλλάξουμε λίγο πορεία και καλωσορίζω όλους ιδιαίτερα στο γεγονός ότι θέτουμε στόχο για την δεύτερη γενιά, αλλά καλό θα ήταν να μην πετάξουμε όλα στα σκουπίδια, όλα εκείνα για τα οποία επενδύσαμε. Ο στόχος για τα σύγχρονα βιοκαύσιμα φαίνεται ότι είναι μετριοπαθής, αλλά θα πρέπει αυτή η νομοθεσία να εφαρμοστεί σε πρώτη φάση. Θα πρέπει να επενδύσουν οι επιχειρήσεις. Το 2020 δεν είναι πολύ μακριά μας και μετά θα έχουμε νέα πρόταση για την περίοδο μετά το 2020 και μετά θα μπορέσουμε να θέσουμε πιο υψηλούς στόχους για τα σύγχρονα βιοκαύσιμα, ελπίζουμε. Να μην ξεχνάμε μετά από όλη αυτή την κριτική ότι τα βιοκαύσιμα πρώτης ή δεύτερης γενιάς και η οδηγία αυτή στο σύνολό της μας βοηθούν να αναξαρτητοποιηθούμε από το πετρέλαιο. Και νομίζω ότι το κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να είναι ενωμένο πίσω από το στόχο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκομφεράτη. Τη μεταρρύθμιση των οδηγιών για την ποιότητα των καυσίμων ή τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια κάνει ένα βήμα προ σωστή κατεύθυνση η Ένωση. Δηλαδή, για αυτό το μέρος του κόσμου να έχει να ετοιμάσει ένα μέλλον πιο πράσινο και βιώσιμο. Σημαντικά αυτούς τους μήνες το, το, το, το Κοινοβούλιο της Πραγματεύσης με αποφασιστικότητα επέλεξε το μεγάλο όραμα για καινοτόμους κανόνες όσον αφορά τα βιοκαύσιμα και υποστήριξε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσης στην καταπολέμηση αλλαγή του κλίματος και την προώθηση της πράσινης οικονομίας. Το κείμενο που απέρασε την Επιτροπή Περιβάλλοντος καθόρισε πρότυπα ακριβώς πάρα πολύ φιλόδοξα τα, η σύναψη της συμφωνίας του Συμβουλίου μειώνει σημαντικά αυτά τα πρότυπα και τα όρια. Παρ' όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Τόρβαλτς για τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε και για τα επιτευθέντα αποτελέσματα. Με αυτούς τους νέους κανόνες παρόλο που έχουν μειωθεί, λέει να σταματήσει επιτέλους ο συναγωνισμός μεταξύ τροφίμων και καυσίμων, λέει η Ευρώπη. Και αυτό είναι σημαντικό. Ε, και θα πρέπει να καταπολεθμεί και η στρέβλωση που αύξησε την τιμή πολλών τροφίμων στις φτωχότερες χώρες για λόγω του μεγαλύτερου κέρδους που δίνουν τα καύσιμα. Άρα ενθαρρύνουμε σωστά τους σωστούς κύκλους και θα μπορέσουμε να τονώσουμε πολλά, σε πολλά κράτη-μέλη σε επενδύσεις που θα οδηγήσουν την ε, στην επίτευξη των στόχων του Κοινοβουλίου για να υλοποιήσουμε αυτό που δεν μπορέσαμε να κάνουμε μέχρι τώρα. Señor Tosenowski. Κύριος Τοσενόσκι. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, η υποστήριξη των κλασικών βιοκαυσίμων αλλά και αυτός ο στόχος του μεριδίου του 10% είναι κάτι το αρνητικό. Θα πρέπει να διορθώσουμε τα κακοσκήμενα. Το 7% επίσης είναι πάρα πολύ υψηλό ως ε, μερίδιο, ως όριο. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε περαιτέρω μειώσει σε εθνικό επίπεδο. Γιατί εγώ διαπιστώνω ότι στη χώρα μου τα βιοκαύσιμα κατέστησαν μια επιχειρήση κερδοφόρα και συνδέθηκαν με ε, κάποιες επιδοτήσεις. Όμως αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι υπάρχει τώρα μια σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, στη χώρα μας ο βασικός παραγωγός βιοκαυσίμων μετέχει στην κυβέρνηση και είναι αυτός ο οποίος ε, δίνει τις επιδοτήσεις. Άρα θα πρέπει να κατέβουμε στο 5-6% και έτσι να αλλάξουν ε, τα πράγματα όπως έχουν σήμερα. Ευχαριστώ κύριο Χάιντεμα, λέει ο πρόεδρος. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε φάνηκε ότι τα βιοκάψιμα είναι αμφιλεγόμενο ζήτημα και αναφέρθηκε ότι πολλά εμπόδια χρειάστηκε να επιπληκτήσουμε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη χρήση των πρώτων υλών. Αυτό είναι και βιώσιμο και οικονομικό. Και εδώ είναι βασικό θέμα οι αγρότες, γιατί παράγουν ε, όλο και πιο πολλά τρόφιμα με πιο πολλή πίεση. Και επιμένουμε λοιπόν στην αποτελεσματική χρήση των πρώτων όρων. Τα βιοκαύσιμα είναι μια ευκαιρία για τους αγρότες και αυτό μπορεί να συνδράμει σε μια κυκλική οικονομία. Χρειαζόμαστε σωστούς και σαφείς στόχους όμως και θα πρέπει να υπάρχει χώρος για πειραματισμό και κοινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Γεωργία έχει τεράστιες δυνατότητες και μπορεί να συμβάλλει στην ε, κοινωνική αυτή ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Σενιόρα Μπόιλαν. Κυρία Μπόιλαν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η τροποποίηση αυτών των δύο οδηγιών μας πήρε πέντε χρόνια. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχασε το Κοινοβούλιο γιατί το Συμβούλιο ήταν ανυποχώρητο. Οπότε τελικά είχαμε μια πολύ πιο απονευρωμένη ρύθμιση από ό,τι θέλαμε. Αυτού του είδους η αλλαγή χρήσης της υγείας τελικά θα έπρεπε να μας οδηγήσει σε καλύτερους στόχους για τα βιοκαύσιμα και ιδίως της πρώτης Και αυτό το 7% που συμφωνήθηκε ε, δεν θα, θα, είναι κάτι καλό για την βιοπικιλότητα και για το περιβάλλον. Αλλά μετά από αυτά τα δύσκολα, τις δύσκολα πέντε χρόνια με τις σκληρές διαπραγματεύσεις θα έπρεπε κάτι καλύτερο να πετύχουμε και να έχουμε κάποιο είδους βιώσιμες μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μόνο η αρχή μιας διαδρομής αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Έχει το λόγο κύριε Χόισλινγκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε την πορεία μας σε ό,τι αφορά τα καύσιμα αυτά, αλλά αυτά που συμφωνήθηκαν δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση, πιστεύω. Πριν από 10 χρόνια είχαμε υψηλές προσδοκίες. Ως εναλλακτική δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες αυτές. Βλέπουμε σήμερα ότι ο κλιματικός ισολογισμός είναι χειρότερος και σε κάποιες περιπτώσεις και από τα ορυκτά καύσιμα. και το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι πράγοντες ILOC πιστεύω ότι είναι σκανδαλώδες. Φυσικά μπορούμε να συζητήσουμε για το κατά πόσον δεν είναι τέλειοι, αλλά το να μην ληφθούν εντελώς υπόψη δεν αποτελεί μια λογική προσέγγιση. Γι' αυτό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συζητήσουμε κατά πόσον μπορούμε απλά να διαγράψουμε τα στοιχεία αυτά. Με το 7% γράφουμε κάτι ως αφή στόχο. Υπάρχει προστασία των επενδύσεων, αλλά είμαστε πάντα πίσω. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν πιστεύω στη δεύτερη γενιά. Το λέω ξεκάθαρα. δεν υπάρχουν ε, αυτά τα υπόλοιπα που ισχυριζόμαστε ότι υπάρχουν και δεν πρόκειται να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι. Θα πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή στην πολιτική μας για την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των μεταφορών. Αυτό αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος Μαζουρώνης. Σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των ε, καυσίμων, θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει στους μελλοντικούς στόχους να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που θα λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες καταστάσεις και τις διαφορετικές συνθήκες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το άνατο σε όλα τα κράτη-μέλη. Η σταθερότητα των ε, της αγοράς θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα εγγυάται. Κατά δεύτερον, προσέγγιση για τις νέες τεχνολογίες. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την απλοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και το κόστος των διακαυσίμων. Αλλά οι τεχνολογίες αυτές είναι σε μία πρώιμη φάση. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει τεχνολογική ανάπτυξη και θα πρέπει να προωθηθεί στο θέμα των βιοκαυσίμων. Μόνο έτσι θα πετύχουμε τους στόχους μας. Tiene usted una tarjeta azul del Σενιόρ Frunzulica. Ο γιος Φρουνθουλίκα έχετε μία μπλε κάρτα. Την αποδέχεστε. Έχετε το λόγο. Η υπερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφό μας, τον κύριο Ματσουλόνης, πώς θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να κινηθεί για να τονώσει την κατανάλωση των βιοκαυσίμων, των προωθημένων βιοκαυσίμων. Ευχαριστώ. Aš manau, kad e, dabar ir, ir, ir apie to, tą dokumentą, kurį mes šnekam, tai ir yra skatinimas ir ieškojimas sprendimų. Το έγγραφο αυτό το οποίο σήμερα εξετάζουμε παρέχει τις ε, απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Αυτό αφενός, αφετέρου. Θα πρέπει να συνενώσουμε και τα συμφέροντα των κρατών μελών, αλλά και τις διάφορες καταστάσεις που επικρατούν, αλλά και τις επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει στον τομέα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε έναν αποδεκτό συμβιβασμό με τους μέγιστους στόχους και τα αποτελέσματα και αφετέρου οι στόχοι θα είναι υψηλοί. Μάλλον, οι θα είναι υψηλή και τα αποτελέσματα πολύ χαμηλά. Το κύριο Μπάλτζο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η οδηγία για το βιοκαύσιμα πέρασε από την φυσιολογική συνήθινη νομοθετική διαδικασία. Όμως Εν προκειμένου, οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου δεν ελήφθησαν υπόψη. Δεν ακούστηκε η φωνή μας. Δείτε λίγο τι λέει το κείμενο του εισηγητή. Και όσον αφορά τα τρόφιμα, αυτό το οποίο κάνουμε είναι προσπαθούμε να επιβάλλουμε κάποιους περιορισμούς στην παραγωγή. Αλλιώς θα υπάρξουν πολλοί δυσάστες συνέπειες στην τιμή των τροφίμων. Θα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό γιατί ήδη σε άλλες υπήρους έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λαβία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύσκολε ήταν οι διαπραγματεύσει, αλλά καταλήξαμε για το άλλο σε κάποια συμφωνία και έτσι έχουμε τώρα έμεση μεταβολή τη χρήση των γιών. Και έχουμε τώρα τον περιορισμό των ε, ε, βλαπτικών εκπομπών ε, που προέρχονται από την καλλιέργεια που οδηγεί στα βιοκαύσιμα. Και θέλουμε τώρα να κάνουμε αυτή την μετάβαση σε κάποια βιοκαύσιμα που να περιορίζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου να έχουμε μείωση των εκπομπών και έτσι αυτό θα γίνει με την έμεση αλλαγή χρήση των γιών και να δούμε ε, πώς θα ε, κάνουν κάποιες αλλαγές στην καλλιέργειά τους ή τώρα ε, ασχολούμενοι με αυτόν τον κλάδο και έτσι θα, αλλάξουν οι οδηγίες που ισχύουν. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τόρβολτς για το έργο του, να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες που συνεργάστηκαν για να εκπονηθεί αυτή η έκθεση αλλά πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον Πρόεδρο της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έτσι καταλήξαμε σε μια συμφωνία για ένα κοινό κείμενο με τη συμφωνία της Κομισιόν. Μπορεί να μην πέρασαν όλες οι λεπτομέρειες που θέλαμε να προωθήσουμε, συγητής και σχεδόν συγητές, αλλά μόνο αυτή η συμβαστική λύση υπήρχε. Δεν είναι δυνατόν, όλα είναι ικανοποιημένοι, αλλά πρόκειται για τον μοναδικό συμβασμό που μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αυτό έχουμε σήμερα αναχειριστεί. Ευχαριστώ πολύ εγώ, λέει ο Πρόεδρος, και το λόγο στον κύριο Λάινεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση για την αναθεώρηση των δύο διών κατέδειξε ότι στο μέλλον θα πρέπει να εστιαστούμε πιο πολύ στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς και κύριε Χόισλινγκ δεν μιλάμε μόνο για όχυρο, άχυρο και για τα υπόλοιπα της γεωργίας, αλλά μιλάμε και για άλλα προϊόντα. Τι κάνουμε λοιπόν για την διερεύνηση αυτές, αυτών των νέων βιοκαυσίμων και την εμπορία τους. Έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα. Θα χρειαστούμε τη βιομάζα για τα αεροπλάνα, για τα φορτηγά, όπου δεν υπάρχουν ακόμα εναλλακτικές. Αλλά σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά οχήματα θα πρέπει να μειωθεί η χρήση τους. Δεν είναι αυτό απαραίτητο γιατί θεωρώ ότι και το υδρογόνο και το ηλεκτρικό αποτελούν άλλες συναλλακτικέ. Και όντως τα βιοκαύσιμα της πρώτης ε, γενιά θα πρέπει να μειωθούν. Εμείς ε, θα θέλαμε 5,5%, 7% προέκυψε. Αυτό θα σημαίνει πιο, πολύ, πιο μεγάλη χρήση γεών. Και γι' αυτό λοιπόν δεν είναι καλό να μην ληφθούν υπόψη τα στοιχεία άλλων. Το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την ε, οδηγία μόνο υπό τον όρο ότι θα, λαμβάνονταν σαν υπόψη, θα εξετάζονταν τα στοιχεία, του όρη του ILOC. Αυτό είναι κακό σημάδι. Κύριε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αυτή η οδηγία έχει σαν στόχο να ξεκινήσει μια πραγματική πολιτική για τα βιοκαύσιμα. Έτσι θα μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μείωση της συμβολής της χρήσης των βιοκαυσίμων μάλλον τη χρήση των βιοκαυσίμων για να μειώσουν τις εκπομπές του θερμοκηπίου. Στην αρχή οι εργασίες εξελίχθηκαν άριστα, όμως το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό. Τα κράτη-μέλη και η βιομηχανία ζήτησε να υπάρχει κοινοποίηση ζήτηση και μάλλον από τις βιομηχανίες να κοινοποιούν για τις εκπομπές τους που συμβάλλουν στα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτό δεν αρκεί. Πολλά κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένες της Πολωνίας θα εφαρμόσουν την οδηγία και θα είναι ε, αβέβαια ποια θα είναι τα συνοδευτικά μέτρα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Σαν πολωνική αντιπροσωπεία ε, θα, θα ψηφίσουμε δεόντως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανάγκη για να αναπτυχθούν και να στηριχθούν οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στον τομέα των μεταφορών είναι σήμερα πιο επιβεβλημένη από ποτέ. Εν τούτης, στην έκθεση που καλόμαστε να ψηφίσουμε για την τροπήση τη σχετική οδηγία, πολλά σημαντικά σημεία απουσιάζουν. Η περαιτέρω αύξηση τη συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια απαιτεί παράλληλε πολιτικέ, την προώθηση δηλαδή κατάλληλων υποδομών, των εξορθολογισμό των καθεστώτων στήριξη, καθώ και την αξιοποίηση των ευκαιριών για διεθνή συνεργασία. επίση είναι πολύ σημαντικό να προσθεθούν μέτρα για τη διασφάλιση τη όθηση των ανανεώσιμων πηγών με το μικρότερο δυνατό κόστο για του καταναλωτέ καθώ και μέτρα στήριξη των μικρών παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. τέλο τα νέα έργα και επενδύσει που χρηματοδοτεί η ευρωπαϊκή ένωση στον τομέα των μεταφορών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος να υποστηρίζουν την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και να προάγουν τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς βεβαίως και μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Πρόεδρο και δεν στον Κύριε Πρόεδρε, στο κόμμα μου δεν έχουμε ιδιαίτερη αγάπη για τα βιοκάψιμα, αλλά ανησυχούμε για το, τη ρυθμιστική αβεβαιότητα που είναι επιζήμια. Είναι ρυθμιστική αβεβαιότητα που δημιούργησε το Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα θεωρήσαμε σαν στόχο να έχουμε 10% βιοκάψιμα. Επιτρέψαμε στη βιομηχανία να κάνει μεγάλε επενδύσει από αυτή τη βάσεω. Μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία επένδυσε μισό δι ευρώ ε, σε, σε αποταστήριο όσον αφορά παραγωγή ελαίου, φινικελαίου. Λοιπόν, τώρα μειώσαμε τα όρια σε 5-6%. Κάνουμε τεράστιε ζημιέ στου επενδυτέ. Του κόβουμε τα πόδια. Δεν μπορεί κανεί έτσι να κάνει να λειτουργήσει μια οικονομία. Γενικότερα βλέπουμε έναν κόσμο που έχει πλημμυρίσει από φθηνό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Και αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί επαρκετών πιστεύω. Οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακο θα αυξάνονται επί δεκαετίε, ανεξάρτητα από αυτά που θα κάνουμε εμεί στο Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, να δώσω μια συμβουλή στου συναδέλφου. Ήρθε η ώρα να συνηθίσουν την ιδέα αυτή. Ευχαριστώ. Κύριε Ροπ, δεν έχω τίποτα να Αλλά χωρίς να το θέλω, σας πέρασα, δεν σας έδωσα το λόγο. Έχετε τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονό ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο σκόπιμα. Τα βιοκαύσιμα πριν από κάποια καιρό φαίνονταν ότι ήταν η καλύτερη λύση για την επίλυση των προβλημάτων μας. Η συμφωνία δε μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τα βιοκαύσιμα και για την δραστική μείωση των βιοκαυσίμων θα δεικνύει άλλη μια φορά ότι θα πρέπει πιο σοβαρά να εξετάζουμε τις αποφάσεις μας. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τις επενδύσεις μας το 2020. Πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν για τα βιοκαύσιμα. και θα πρέπει να ε, εξετάσουμε και τα θέματα αλλαγής χρήσης γεών και να δημιουργήσουμε τους όρους για τη νέα εκμετάλλευση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πράγματι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα πάρα πολύ επίμαχο και επί σειρά ετών το πολεμούσαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τα πάντα για να προωθήσει την ανάπτυξη βιοκαυσίμων και εν συνεχεία τι διαπιστώσαμε, ε, απογοητευτήκαμε. Όλα αυτά αμφισβητήθηκαν. Τελικά αυτή η συμφωνία ίσως δεν είναι αρκετά φιλόδοξη για κάποιους, ίσως θα ανησυχεί άλλους. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ισορροπημένη και ότι επιτρέπει να διατηρήσουμε τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν για τα βιοκαύσιμα της πρώτης γενιάς. Ταυτόχρονα όμως φροντίζει ούτως ώστε αυτά τα βιοκαύσιμα να μην μπουν σε ανταγωνισμό με την παραγωγή τροφίμων και να μην παράγουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε υπερβολικό βαθμό. Λοιπόν, οι επενδυτές δεν θα μπορούσαν να είναι θύματα μιας ισοσπαστικής αλλαγής πολιτικής. Τους χρειάζεται χρόνος όταν επενδύουν. Πρέπει να υπάρχει μακροπρόθεσμο όραμα στον αφορά την προσέγγιση μας. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα, ε, θα Θεωρώ ότι είναι αβέβαιοι υπολογισμοί που έγιναν για το αντίκτυπο και αμφισβητήσιμη μέθοδοι επιστημονικά όσον αφορά την, ε, πώς επιδρούμε στη χρήση των γεών. Αυτή η ε, συμφωνία επιτρέπει κάποια ε, δυνατότητα ενημέρωσης εν αναμονής βελτίωση των υπολογισμών. Λοιπόν, ο στόχο που έχουμε θέσει για το 0,5% των καυσίμων είναι ρεαλιστικό στόχο, αλλά λυπούμε διότι δεν είναι περιοριστικό. Διότι οι πόροι είναι πολύ λίγοι για την παραγωγή αυτών των καυσίμων. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί τεχνολογικά από τα βιώσιμα καύσιμα και γι' αυτό σίγουρα θα πρέπει να υποστηρίξουμε την έρευνα και ανάπτυξη στον συγκεκριμένο τομέα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Παχνιού έχει το λόγο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Επιτέλους στάσαμε στο, τέλμα, στο τέλος αυτής της ε, για τα βιοκαύσιμα της πρώτης γενιάς. Ήταν ελκυστική αρχικά η όλη να μειώσουμε τη χρήση του πετρελαίου. Δυστυχώς ε, ε, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Ε, αποφάσισε όμως να γυρίσει την πλάτη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα καύσιμα που μόνο κατά όνομα είναι βίο ε, θέλαμε να, να είναι περιοριστικό ο συμβιβασμό. Θέλαμε να πετύχουμε στο, στην COP21 στο Παρίσι να έχουμε συμφωνία. Τώρα στέλνουμε ένα θετικό μήνυμα πλευρά Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε σοβαρά, να προσπαθήσουμε να έχουμε ε, μια οικονομία που δεν θα παράγει πολύ άνθρακα. Αλλά πόρα απέχουμε από το τέλειο θα ήθελα να προχωρήσουμε περισσότερο, ζητώντας να συμπεριληφθούν ε, και άλλα κριτήρια στην βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων επιβάλλοντας περιοριστικούς στόχους για τα βιοκάψιμα θα είναι ένας συμβιβασμός που είναι ένα βήμα σημαντικό. Ένα βήμα όμως, έχουμε κάποιο όριο, το μέλλον ανήκει στα προθυμένα βιοκαύσιμα, περνώντας από τα βιοκαύσιμα της πρώτης γενιάς. Λοιπόν, το βασικό το έχουμε. Η Ευρώπη αναγνωρίζει επιτέλους ότι τα βιοκαύσιμα ε, τα, από υγειοργικά δεν είναι μια απάντηση στην αλλαγή του κλίματος. Τα κράτη-μέλη, ξεκινώντας και από τη Γαλλία, πρέπει να θέσουν στόχους μέχρι το 2020 να δημιουργήσουν 100 με 150.000 θέσεις εργασίας στον τομέα των προθυμένων βιοκαυσίμων. Πιστεύω ότι έχουμε πρόκληση μπροστά μας. Θα την αντιμετωπίσουμε στην COP21 το Δεκέμβριο στο Παρίσι. Και αυτή η απόφαση που θα λάβουμε σήμερα πιστεύω ότι ακολουθεί σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Γκέρλινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον ε, εισηγητή. Πρόκειται με μεγάλη διαδρομή που ξεκίνησε από την προηγούμενη θητεία. Τώρα νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέρμα και είναι εντυπωσιακό ότι εδώ κανένα δεν φαίνεται να θέλει να λάβει ευθύνη για την συμφωνία ή τη συμφωνία του 2008 για το όριο του 10%. Ξαφνικά φαίνεται σε όλους ε, κάτι το πάρα πολύ κακό. Κι όμω. εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογη τη συμφωνία γιατί το πρώτο το οποίο προγύπτει είναι ότι έτσι ελκύσαμε το ενδιαφέρον των επενδυτών. Οπότε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο αν θέλουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα που να είναι πιο μακρόπνο θα πρέπει να προσπαθήσουμε και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να μην δυναμητήσουμε αυτό που πετύχαμε τώρα λίγο πριν από το τέρμα τη διαδρομής. αυτό το 7% δεν είναι κακό. Πάρα πολύ σήμερα το πρωί είπαν ότι πέρασε θέση του το Συμβούλιο, εγώ θεωρώ ότι είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο πετύχαμε και όσον αφορά το καύσιμο αυτό γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε πότε η επιστήμη θα μπορεί να ελέγξει το προϊόν κάτι το οποίο δεν ισχύει ακόμη και για τις διαπραγματεύσεις ε, που βγάζω το καπέλο μου στον κύριο Τόρβελτς αλλά είναι αλήθεια ότι αυτό που θα μπορούσε να ισχύει είναι να έχουμε ένα δεσμευτικό στόχο για το βιοκαύσιμο. Δεν το πετύχαμε αυτό. Αυτό ήταν ο στόχο που ήθελαν όλε οι πολιτικέ ομάδες σε όλο το φάσμα του Κοινοβουλίου. Δεν το πετύχαμε αυτό. Οπότε νομίζω θα πρέπει να ντρέπονται οι διαπραγματευτέ γιατί δεν πέτυχαν αυτό το οποίο όλοι θέλαν. Κύριο Μαχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, έκανα μια τροπολογία για τη μείωση του φάσματος το, του ορίου μάλλον των παραδοσιακών διακαυσίμων στο 6% και αν ήταν δυνατόν θα ήθελα να προτείνω πλήρη διαγραφή της, της οδηγίας αυτής γιατί πρόκειται για ένα τρατούργημα οδηγεί σε αύξηση τιμών σε πείνα σε πολλές χώρες του κόσμου πρόκειται για ένα σύστημα όπου ολιγάρχες επωφελούνται και προτίζουν και στη Τσεχία ο κ. Μπάμπης, ένας από αυτούς τους ολιγάρχες, εξαγόρασε καταρχάς τους πολιτικούς για να επιτρέψει το έλεο κράμβης να συνεχίσει να καλλιεργείται και μετά αγόρασε τα μέσα ένα κανάλι, σε, μπήκε μέσα στον τύπο, έγινε πολιτικός, πήρε υψηλόμαθμες θέσεις και τουλάχιστον ε, ας περιορίσουμε το όριο των ε, παραδοσιακών ε, βιοκαυσίμου στο 6%. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάμε. Είναι θετικό το αποτέλεσμα. Ήμουν ε, εκπρόσωπο τη ομάδα μου το 2009 και τότε οι πράσινοι μα έλεγαν κι άλλο κι άλλο. Τώρα λοιπόν θέλουν ε, μεταστροφή. Να σκεφτούμε την προστασία όμω των επενδυτών. Κλείνει όμω το μικρόφωνο του κ. Λάνα. Εκτό μικροφώνου. I need to start. Ah, Good. Good is better. So. Μάλιστα, πολύ καλύτερα. Πολύ ωραία. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο του Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο από ό,τι το παρουσίασα. Είναι μια σωστή μέση οδό μεταξύ προστασία επενδυτών και των απαιτήσεων που τίθενται από το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερως από τους Πρασίνους το 2008. Τότε ήμουν λοιπόν εκπρόσωπο τη ομάδα μου και τότε μας έλεγαν κι άλλο. Πιο υψηλέ αξίες. Και τότε ξέραμε ποια ήταν τα αποτελέσματα των βιοκαυσίμων. Τώρα δηλαδή μία ναι, μία όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλό ο συμβιβασμό. Το αποτέλεσμα είναι καλό. Ο, οι στόχοι τη Επιτροπή Βιομηχανία, όπω αποφασίστηκαν από την ε, Επιτροπή Ήτρε, ακολουθήθηκαν σε μεγάλο βαθμό πολλές επιστημονικές, ε, επιστημονικά τεκμήρια ε, μας οδήγησαν στα αποτελέσματα όπως το reporting, ένα πρώτο βήμα, το 7% αποτελεί καλό βήμα, ακόμα και αν είναι πιο ψηλό ποσοστό από αυτό που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Τα συμβατικά βιοκαύσιμα έχουν ε, μια προστασία και ασφάλεια. Το 0,4% για τη δεύτερη γενιά δεν είναι αρκετά φιλόδοξο και είναι Λυπηρό το ότι δεν υπάρχει κάτι ξεχωριστό κατά την όλοι. Θετικό είναι το ότι αποφασίστηκε να συνεχιστεί μετά το 2020. Θετικό λοιπόν είναι ο συμβιβασμό μεταξύ σταθεροποίηση αγορά, μείωση τη εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα. Και τώρα θα πρέπει να δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει από το 2020 και μετά. Ε, εσείς έχετε λοιπόν πλέον το λόγο να καταθέσετε μια νέα πρόταση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάντεμπαχ. Η κυρία Καντεμπάχ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ένας συμβιβασμό μπορεί να εγκριθεί ή να θεωρείται αποδεκτός. Ε, για μένα είναι ίσα ίσα αποδεκτός, είναι καλύτερα από αυτό που είχαμε προηγουμένως. Συχνά με ρωτάνε γιατί είσαι κατά των βιοκαυσίμων, τόσο καλά ακούγονται. Νομίζω ότι πολλοί ήμασταν πεπισμένοι ότι είχαμε αποφασίσει κάτι θετικό, αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι στην πραγματικότητα υπήρξε μια μετεγκατάσταση από μια παραγωγή για τα ανθρώπινα τρόφιμα και στις ζωοτροφές ε, σε μια παραγωγή για να γεμίζουν οι δεξαμενές. Το βιοσπρίτ, το αγροσπρίτ δεν ήταν αυτό που θέλαμε τελικά άλλαξε η αλλαγή της χρήσης ε, γεών, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε τρίτες ε, χώρες. Και τελικά, αυτά που πριν από 10 χρόνια αποφασίσαμε με καλές προθέσεις, τελικά να έχουν τους αντίθετους στόχους, τους αντίθετο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είναι αποδεκτός ο συμβιβασμός. Συχνά ακούσαμε, σε πολλές περιπτώσεις ακούσαμε σήμερα ότι θα πρέπει να υπάρχει και προστασία των επενδύσεων. Αυτή η προστασία θεωρώ στο 7% είναι πολύ μεγάλη. Για το 6% θα θεωρούσα πιο σωστό συμβιβασμό. Ακούσαμε επίσης ε, από διάφορους σήμερα ότι θα συνεχιστεί αυτή η παραγωγή, ότι θα υπάρξει μια πιο προοδευτική παραγωγή και θα πρέπει να κοιτάξουμε το πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την κινητικότητα με την πιο χαμηλή επιβάρυνση. Αυτό χρειάζεται για το μέλλον η Ευρώπη. Κυρία Αγίου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε και αγαπητοί συνάδελφοι. Το πρώτο που πρέπει να κάνω είναι να συγχαρώ τον εισηγητή, την Λετωνική Προεδρία αλλά και την Επιτροπή για τα αποτελέσματα που απέσπασαν και αυτή τη δύσκολη συμφωνία. Το να προωθήσουμε αυτά τα προωθημένα βιοκάψιμα και κλείνουμε την πόρτα με αυτόν τον τρόπο στην προηγούμενη γενιά. Αυτό ήταν ένας στόχος που ήταν λογικός. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για την πρώτη οδηγία για βιοκαύσιμα και θυμάμαι με τι ενθουσιασμό υποδέχθηκαν οι πράσινοι α, τους δεσμευτικούς προωθημένους στόχους. Όμως όλοι δικαιούμεθα να αλλάξουμε γνώμη. Νέες τεχνολογίες για μείωση των εκπομπών τώρα, ούτως ώστε να έχουμε ε, μια προστασία επαρκή. Αυτό γίνεται με τα βιοκαύσιμα και έχουμε ποιοτικέ μεγάλες επενδύσεις. Και τώρα θα αντικαταστήσουμε ένα, μια μεγάλη μερίδα των ε, ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές. Θα πρέπει να κάνουμε καμία αξιολόγηση. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και θέλουμε από τη θεωρία να περάσουμε στην πράξη, χωρίς όμως να τηρούμε κάποιες προϋποθέσεις. Άρα θα πρέπει τα κρατη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Και έτσι να δούμε το πώς τα βιοκαύσιμα να έχουν όλο ένα και μεγαλύτερο μερίδιο σε νέες πηγές ενέργειας στις μεταφορές μέχρι το 2020. Ευχαριστούμε λέει και ο Πρόεδρος και δίνει το λόγο στον κύριο Ποκ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σήμερα ψηφίζουμε μια πρόταση η οποία δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ε, του Κοινοβουλίου για την πολιτική βιοκαυσίμων, ούτε ανταποκρίνεται στις αρχικές ιδέες του Ευρωπαϊκού Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνονται τι προσδοκίες κάποιων κρατών μελών και στις προσδοκίες κάποιου τομέα της βιομηχανίας αυτά τα κράτη-μέλη. Δεν εκπλήσωμε που το Συμβούλιο δεν εκπροσωπείται καν εδώ σήμερα, διότι θα έπρεπε να παραδεχτεί ότι το Συμβούλιο στηρίζει ένα δημοκρατικό έλλειμμα. Δύο τρίτα των βιοκαυσίμων στην αγορά αποτελείται από καύσιμα πρώτης γενιάς και οι δραστηριότητες των παραγωγών αυτών έχουν γίνει αισθητέ ε, στο Συμβούλιο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει πολλά περισσότερα, θα μπορούσαμε να είχαμε ακούσει την καινοτόμα βιομηχανία, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και αντί να σταματήσουμε δεχτήσουμε την αύξηση χρήσεως καυσίμων της πρώτης γενιάς, δεχθήκαμε την αύξηση της χρήσεως αυτών με τις παρενέργειες που συνεπάγεται αντί να στηρίξουμε ε, την καινοτομία και τη βελτίωση. Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα είναι καλύτερα από το status quo και καταψήφιση της προτάσεως θα σήμαινε την παραμονή του status quo. Έχουμε σωστά όρια τα βιοκαύσιμα και για τη σωστή χρήση των γεών και στηρίζουμε και κάποιες καινοτομίες. Στέλνουμε στο Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη ε, πολύ άσχημο μήνυμα θα στείλουμε μάλλον αν ε, τελικά πετύχουμε συμβιβασμό ο οποίος δεν είναι ο σωστός. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βυσίτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η λύση που υιοθετήθηκε το 2008 μας δείχνει σαν να βλέπουμε σε καθρέφτη το πώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες. Ποια είναι τα αποτελέσματα. Τα είδαμε. Εγκαταλείπουμε τον το στόχο του 10% που θεωρήσαμε ότι μπορεί να διατηρηθεί τότε. Ήταν προφανής επιλογή τότε. Έγιναν επενδύσεις, πήραν κάποιοι πιστώσεις για να επενδύσουν. Αναφέρομαι σε χώρες που επένδυσαν στα βιοκαύσιμα που καλλιεργούνται στην Ευρώπη. Δεν μιλάω για παραγωγή καυσίμων από το φινικέλαιο παραδείγματος χάρη. Αναφέρομαι στη χώρα μου όπου έχουμε εκατομμύρια τόνων καυσίμων που έχουν παραχθεί τοπικά σε εμά. Και δεν μιλώ για εισαγόμενο φινικέλαιο θα πρέπει να βασιστούμε σε σωστά επιχειρήματα και στην κοινή λογική στις λύσεις που θα βρούμε όσον αφορά τα ενεργειακά ζητήματα. κοιτάξτε, ρίχνουμε στα σκουπίδια το 1 τρίτο των τροφίμων που παράγονται. Πολύ συχνά έχουμε τέτοια απόβλητα τρόφιμα. 10 ε, εκατομμύρια τόνους τροφίμων πετάμε που έχουν παραχθεί κάπου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο τα βιοκαύσιμα μας εμποδίζουν από την πλήρη χρήση των τροφίμων. Ποια ενέργεια είναι καλύτερη, η ενέργεια εκείνη που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, αυτή που έχουμε πετάξει στα σκουπίδια. Ας προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε πολιτική τέτοια που θα μας επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά δεν χρειαζόμαστε και την έγκριση μέσα επανάσταση τώρα, διότι ήδη έχουν γίνει επενδύσεις. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ο Σωρίνιο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή η οδηγία χρονολογείται από μια περίοδο πριν από την ανακοίνωση για την Ενεργειακή ε, Ένωση. Μπορούμε να προβούμε σε μια επαναξιολόγηση με την ενόψη νέας προοπτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθεί ε, την ασφαλή εφοδιασμό στην ενέργεια, ενεργειακή απόδοση, καινοτομία, έρευνα, χρήση νέων καυσίμων. Οι προτάσεις της ε, εκθέσεως είναι καλά ισορροπημένες εν γέννη καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξη πρόταση για την πρόθεση και χρήση ανανοσίμων πηγών ενέργειας στον μεταφορικό τομέα ε, μέχρι το 2020. Σε αυτό το πλαίσιο προχωρούμε πέρα από τα κίνητρα για τη χρήση προθυμένων τεχνολογίων για καύσιμα νέα γενιά χάρη που μειώνουν τον ανταγωνισμό με άλλου τομεί όπω είναι η παραγωγή των τροφίμων και ε, μειώνουμε έτσι την παραγωγή των αερίων του θερμοκηπίου. Θέλουμε φιλόδοξο στόχο για την ηλεκτρική κινητικότητα, Φερρυπίν. Η ηλεκτρική κινητικότητα μπορεί να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπορεί να συνεργαστεί με τα βιοκαύσιμα και να έχουμε υψηλά επίπεδα τοπικά παραγόμενης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών και μπορούμε να πετύχουμε ασφαλή φουδιασμό ενέργεια, να μειώσουμε την εξάρτηση και να είναι στην πρώτη γραμμή Ευρωπαϊκή Ένωση με νέας εποχής για τον τομέα των μεταφορών. Αυτό που κάνουμε μέχρι το 2020 θα οδηγήσει θα αφήσει σφραγίδα όσον αφορά την μελλοντική μας δυνατότητα να ηγηθούμε στην αλλαγή στο μεταφορικό τομέα. Και ο πλανήτης χρειάζεται μια φιλόδοξη Ευρώπη. Το έγγραφο που έχουμε μπροστά μας σήμερα επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει θετικά προς την επίτευξη του στόχου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλετ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Θα ήθελα να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που μετά από πολλά χρόνια διαπραγματεύσει έχουμε μια συμφωνία. Η συμφωνία το ξέρουμε, δεν είναι τέλεια. Και θα πρέπει να περάσουμε οριστικά στο μονοπάτι των προηγμένων βιοκαυσίμων που δεν ε, επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν αυξάνουν τις τιμές των τροφίμων. Οι παραγωγοί λοιπόν ξέρουν σήμερα που βρίσκονται και μπορούν να προγραμματίσουν τις επενδύσεις τους με την παραγωγή των προηγουμένων βιοκαυσίμων. Και η συμφωνία αυτή προφανώς δεν είναι σαφήνεια για τους παραγωγούς παραδοσιακών βιοκαυσίμων. Έχουν χρόνο να προετοιμαστούν και να περάσουν στην παραγωγή των προηγμένων ε, διακαυσίμων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Και τέλος, συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι που με την συμφωνία αυτή κάνουμε μία πρώτη προσέγγιση για την ηλεκτρική οδήγηση πάντα βάσει ανανεώσιμων πηγών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι που κάνουμε ένα πρώτο βήμα και ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα για τον πυλώνα της Ενεργειακής Ένωσης που έχει ανακοινώσει η Επιτροπή ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μετά από αυτέ τι σκληρέ συζητήσει όσον αφορά το μέλλον των ε, βιοκαυσίμων στην Ευρώπη, το Κοινοβούλιο τελικά σπέβδει να ψηφίσει αυτό το κείμενο που θα στείλει αυτό το σημαντικό μήνυμα όσον αφορά την, ε, τον αγώνα μας για την προστασία του κλίματος και της οικονομίας οπότε τώρα θα μπορέσουμε να δούμε τι έχει επιτευχθεί όσον αφορά την παραγωγή των βιοκαυσίμων ε, που ονομάζονται παραδοσιακά, που προέρχονται από την καλλιέργεια κάποιων ε, τροφίμων γεωργικών καλλιεργειών και θα πρέπει να αλλάξει η χρήση της γης και όμως να μην καταλαβούν τα δάση και αυξηθεί το διοξείδιο του άνθρακος που εκπέμπεται τώρα. Ε, έχουμε την πρόταση του Συμβουλίου, θέλαμε να δούμε ποια είναι η καλύτερη συμφωνία, να γίνει ένα βήμα προς το εμπρός για να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Έχουμε αυτή την ε, πρόκληση και θέλουμε να ε, ισχυροποιηθεί η θέση μας ως Ευρώπη για την αλλαγή του κλίματος πράσινη οικονομία με κάποιες ε, πολιτικές δίκαιες και βιώσιμες. Ε, Βιωσιμότητα για την προστασία του περιβάλλοντος, έξοδος από την ε, κρίση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Λίνς. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εκείνους που αντιμετώπισαν το πρόβλημα αυτό μετά από πολλά χρόνια αμφιλεγόμενων συζητήσεων κατάφεραν να πετύχουν ένα συμβιβασμό. Είμαι ικανοποιημένο που έχουμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο πλέον και πιστεύω ότι συνολικά πρόκειται για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Τα βιοκαύσιμα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό σε μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας και στη μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ε, Επίση υποστηρίζουν την ενεργειακή μας ανεξαρτησία. Τα βιοκαύσιμα πρώτη γενιά. Θεωρώ ότι εδώ πετύχαμε έναν ε, καλό συμβιβασμό. Είναι πολιτική, πολιτικό το θέμα. Οι αποφάσεις μας να είναι βιώσιμες. Χρειάζεται ε, ασφαλεία προγραμματισμού, προστασία των επενδύσεων. Το γεγονός ότι Ελήφθησαν υπόψη στις εκθέσεις τα σχόλια του, τα παράγοντες του Άιλο, αλλά δεν ε, μπήκαν στο τελικό κείμενο. Θεωρώ ότι είναι μια καλή απόφαση με την προηγούμενη έκθεση. Θέσαμε το μονοπάτι για το μέλλον, τα βιοκαύσιμα είναι σημαντικά, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τι θα γίνει και να προσθέσουμε ιδιαίτερα τις ευαίσθητες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Κούμπουλα Νάτρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την βιοοικονομία ήμουν πρόεδρος στη σχετικά ομάδα εργασία τότε και είμαι ικανοποιημένη που καταφέραμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό επί του οποίο μπορούμε να ψηφίσουμε. Στόχο θα πρέπει να είναι να κοιτάξουμε τι θα γίνει μετά το 2020 γιατί το έτος αυτό θα έρθει σύντομα. Θα πρέπει λοιπόν να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα στις μεταφορές χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός με την ε, βιομηχανία των τροφίμων. Για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δάση και τα σοκομεία της Βόρειας Ευρώπης με τέτοιο τρόπο ώστε το ξύλο να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο και έτσι να μειωθούν και οι εκπομπές. Δυστυχώς η σημερινή πρόταση δεν δίνει μεγάλη σιγουριά στον κλάδο για το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον, το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν λυπάμαι που δεν υπάρχουν και δεσμευτικοί στόχοι. Υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια για τα εθνικά κράτη-μέλη. Στη Φιλανδία 10% ε, ο στόχος του 10% σε μείωση των εκπομπών έχει επιτευχθεί. Είναι βέβαιη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει σωστή ιστορική αγορά για τα βιοκαύσιμα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κιόστινγκερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και να συμφωνήσω με όσους δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με το συμβιβασμό αυτό. Φοβάμαι ότι η συζήτηση αυτή γίνεται μόνο σε ιδεολογικό επίπεδο ουσιαστικά. Και αυτό στην πλάτη των παραγωγών στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει βεβαιότητα και ασφάλεια για τους παραγωγούς. Το αποτέλεσμα που θα ψηφίσουμε είναι αποδεκτό, αλλά σίγουρα δεν επαρκεί. Ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αποτελεί. Και αυτό μόνο. Η βιεθανόλη και το βιοδίζελ θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζονται. Και είναι η μονοδιάστατη συζήτηση. Στην Αυστρία η παραγωγή βιοεθανόλης και των παραπροϊόντων είναι ένα σημαντικό θέμα 100% ε, ελεύθερο από γενετικά τέτοια ζητήματα και όσον αφορά τους ε, όρους του Άιλο ευτυχώς δεν συμπεριλήφθησαν γιατί είναι πολύ αμφισβητούμενα από πλευράς επιστημονικής και να συμφωνήσω με την προηγούμενη μιλήτρια που είπε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει και μετά το 2020. Θα χρειαστούμε σημαντικά μέτρα για τη μείωση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και του καθεξής. Σημαντικό είναι να συνεχίσει η πρόθεση των βιοκαυσίμων απορρίμματα, σπέρι κτλ. Όλα αυτά αποτελούν το μέλλον των βιοκαυσίμων. Κύριε Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Με μεγάλη μου χαρά να σας μιλήσω πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα. Όταν ε, ανα, αναλάβετε τα καθηγοντά σας υποσχεθήκατε να υπάρχει μια γενική πολιτική για να σταματήσουμε να είμαστε τόσο χαιρετημένοι από τα ορυκτά καύσιμα και να έχουμε τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε βεβαίω και εδώ πέρα έχουν σημασία τα βιοκαύσιμα, ιδίω όσον αφορά τι μεταφορέ. Θα πρέπει να δεχτούμε ότι δεν έχουμε ε, λάβει τα σωστά μέτρα για μείωση των εκπομπών. Έχουμε ε, τη δεδομένη οικονομία μα, όπου έχουμε όλα αυτά τα φορτηγά, ε, τι νταλίκε, τα αυτοκίνητα στου δρόμου. Οπότε και όπω είναι του είναι εύστοχο ο συμβασμό, διότι τώρα έχουμε αυτή τη σωστή ισορροπία μεταξύ πρώτης και δεύτερης γενιάς των βιοκαυσίμων και επομένως τα προηγμένα βιοκαύσιμα είναι το μέλλον. Συμφωνούμε με αυτή τη ρύθμιση. Επίσης ε, θα μειωθούν τα, οι αρνητικέ συνέπειες, θα ελκύσουμε τους επενδυτές. Είναι αυτό το οποίο θα πρέπει ε, να, κάνουμε αυτό αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο μέλλον. Επίση, έχω μιλήσει με πολλούς τέτοιους επενδυτές που λένε ότι ήταν μεγάλη απώλεια ευκαιρία στο να μην χρησιμοποιηθεί ε, τα σκουπίδια για αυτό το λόγο στο παρελθόν και να μην έχει υπάρξει κάποια λύση όπως τώρα στο παρελθόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Πρόεδρος. Και τώρα, αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση γιατί προχωρούμε στη διαδικασία Catch VI και όσοι λάβουν τον λόγο θα έχουν ένα λεπτό στη θέση τους. Κύριε Μπόβικ, έχει το λόγο. E, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στηρίζω τη συμβιβαστική αυτή η πρόταση. Πρόκειται περί απαντήσεως στο πρόβλημα που προέκυψε λόγω των πολύ φιλόδοξων στόχων που είχαμε θέσει. Είχαμε αρνητικές συνέπειες λόγω του ILUC. Τα τρόφιμα γινόταν όλο και πιο ακριβά. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω. Σκεπτόμενοι την Ενεργειακή Ένωση και την όλη έννοια της ενέργειας, θα πρέπει να διευκολύνουμε την επίτευξη του καθοριστέντος στόχου. Θα πρέπει να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Αυτό είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Στον μεταφορικό τομέα έχουμε τις περισσότερες δυνατότητες να το πετύχουμε αυτό. Έχουμε προβλήματα με τους τεθέντε στόχους και από την τεχνολογική πλευρά. Αυτή η πρόταση θα μας οδηγήσει σε μια βελτίωση στον τομέα των τεχνολογικών εξελίξεων. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Εάν προχωρήσουμε σημαντικά εκεί, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πετύχει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι ο σωστός δρόμος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ καταρχάς τον εισηγητή, παρόλο που καμιά φορά έχω το αίσθημα που δεν είναι ικανοποιημένο με το αποτέλεσμα που πέτυχε. Πριν όμως ψηφίσουμε μια έκθεση θα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει να μην την ψηφίσουμε. Είναι ένα πολύ περίπλοκο και ευαίσθητο πρόβλημα αυτό που συζητούμε και δεν μπορεί να οδηγήσει σε συμβιβασμό που ικανοποιεί όλους από την πλευρά μου πιστεύω ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε λιγότερο μια βάση πολιτικής θέσεως, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε βάση τη λογική και να σκεφτούμε τους ε, συμπολίτες μας. Είναι ένα βήμα σημαντικό αυτό θα πρέπει να γίνουν σωστές επενδύσεις στο μέλλον και γι' αυτό κύριε Επίτροπε θα πρέπει να πείσετε τους συναδέλφους σας στο Κολέγιο των Επιτρόπων να δώσουν περισσότερα χρήματα στην έρευνα διότι η πρόοδος βασίζεται στην έρευνα. Το σωστό ενεργειακό μείγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να δούμε και, ποιες, και πώς το ενεργειακό κόστος επηρεάζει τους ε, συμπολίτες μας. Έχουν δικαίωμα όμως και σε ένα καθαρό περιβάλλον, πρέπει των πτυχών. Ε, αυτών. Ο συμβιβασμό είναι σημαντικό βήμα, αλλά δεν έχουμε λύσει τα πάντα μέσω του συμβιβασμού. Μπορούμε να πούμε ότι σημειώθηκε μια πρόοδο και μπορούμε να το δείξουμε αυτό στου συμπολίτε μα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μαριά νομίζω ότι δεν είναι εδώ. Ο κύριος Τζάκοβιτς λοιπόν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευτή εξ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι Υποστηρίζω απόλυτα την έκθεση αυτή. Και αυτό γιατί γνωρίζω ότι ο Κριστόρ Βάλς, ο εισηγητής, έκανε τα πάντα, ό,τι περνούσε από το χέρι του για να πετύχει τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό. Και να ληφθούν οι υπόψεις στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και οι θέσεις του Κοινοβουλίου. Εγώ προσωπικά ε, ήμουν σε θέση να κάνω διάφορα πράγματα που ήταν σημαντικά για την έκθεση. Αλλά πρέπει να πω ότι τότε δεν έκανα πολλά όταν ε, μιλήσαμε για την, ε, τα δύο πρώτης γενιάς. Θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να προσανατολιστούμε προς την κατεύθυνση αυτή και καλό τους πάντες ε, να επενδύσουν προκειμένου όλα τα απορρίμματα να μπορέσουν να αποτελέσουν αποτελεσματικά. Ο κύριο Κλέζος. Ε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα βιοκαύσιμα πέρα από τη μόλυνση του περιβάλλοντος την οποία συνεπιφέρουν με τη, κυρίως από το διοξίδιο του άνθρακα συντελούν στην αύξηση της θερμότητας της γης. Αυτή η αύξηση της θερμότητας δημιουργεί δύο φαινόμενα. Λιώνουν οι πάγοι. Εκεί που λιώνουν οι πάγοι ανεβαίνει ο φλοιός στο σημείο αυτό όπως έχουμε καταμετρήσει στην Γρυλανδία και όπως έγινε και στα Ιμαλάια και γι' αυτό έγινε ο μεγάλος σεισμός των Ιμαλαίων. Το δεύτερο φαινόμενο είναι ότι με το λιώσιμο των πάγων δημιουργείται τεράστια αύξηση της εξάτμισης και της εξάτμισης με αποτέλεσμα να έχουμε ρόχο να έχουμε πλημμύρες και να έχουμε κατάκληση των εδαφών στα χαμηλά σημεία. Πέρα από αυτό όμως το σημείο δημιουργείται ένα τεράστιο βάρος που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις συνέπειες. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου κρούω τον κόδωνα του κινδύνου εάν δεν πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ο κύριος Τούρμες. Σας ευχαριστώ. Ως πρώην εισηγητής ε, ήθελα να δω ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Συνολικά δεν θεωρώ ότι είναι πολύ καλό συμβιβασμό. Είναι μάλλον αδύναμος. Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το Κοινοβούλιο όσο με την άποψη του Συμβουλίου. Θα πρέπει θα πρέπει να περιοριστεί η πρώτη γενιά των βιοκαυσίμων. Έχουμε υπερβολικά μεγάλο ανταγωνισμό με τα τρόφιμα. Το 7% είναι πολύ υψηλό, ίσω υπερβολικά υψηλό, αλλά τι να γίνει. Κατά δεύτερον, χρειάζεται μια μεθοδολογία για υπάρξει ισοσκελισμός όλου του, του, των εκπομπών διοξιδίου του ανθρακά των βιοκαυσίμων. Και κατά τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσεί, ε, Επιτροπή Καλνιέτε, καλείστε να ε, δώσετε την ασφάλεια των ε, επενδύσεων. Αφού το 0,5% για το δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων θα πρέπει λοιπόν μετά το ισχνό αυτό συμβιβασμό να κάνει η Ευρωπαϊκή Πολιτική μια έρευνα για να δει τι μπορεί να δαπανίσει στην έρευνα, στις επενδύσεις, Βουλγαρία, Πολωνία, Ουκρανία, ενδεχομένω να χρειάζονται επενδύσεις για αυτή τη δεύτερη και τρίτη γενιά βιοκαύσιμα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους τους ε, βουλευτές για τα όσα είπαν σε αυτή την ε, συζήτηση. Ακούσαμε όλα αυτά τα επιχειρήματα και η συζήτηση αυτή ανέδειξε το πόσες δυσκολίες ανέκυψαν κατά τις διαπραγματεύσεις για αυτή την οδηγία και τελικά ο συμβόλος και όπως είπατε και εσείς δεν ικανοποιούνται 100% όλοι ή κανένας χωριστά όμως με το τελικό αποτέλεσμα έχουμε τώρα αλλαγή της χρήσης της γης και δυνατότητα για προηγμένα βιοκαύσιμα. Για να δούμε τώρα τι έγινε και ποιο είναι το γενικότερο πλαίσιο. Έχουμε αυτή την ε, στρατηγική και αυτό αντιστοιχεί στην ιδέα του Προέδρου Γιούνκερ, ούτως ώστε να είμαστε πρωτοπόροι ως Ευρωπαίοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όμως, για αυτή τη νέα πολιτική θα κάνουμε μία μετάβαση. Θα αφήσουμε πίσω αυτό το οικονομικό μοντέλο που στηρίζεται στα ορυκτά καύσιμα. Τώρα όμως θα έχουμε τα προηγμένα θα αφήσουμε πίσω μα τις απαρχαιωμένε μορφές παραγωγής και ενέργεια. Έχουμε τώρα αυτή την καλλιέργεια ε, γεωργικών προϊόντων, έχουμε το iLook, όλα αυτά θα διαμορφώσουν τη στρατηγική μας. Το δε, ε, ο δε χάρτης πορείας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μα οδηγήσει ε, με αυτά τα μέτρα στι ανέσμε πηγέ ενέργεια. Θα έχουμε τα βιοκαύσιμα που θα κυριαρχήσουν μετά το 2020. Όπως είπατε και εσείς, διαμορφώθηκε αυτή η δέσμη μέτρων. Να πάμε σε ολοκληρωμένη πολιτική και να εκμεταλλευτούμε την πείρα την οποία αποκτήσαμε σε αυτή τη διαδρομή για το θέμα. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Τόρβαλς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Κανιέτα. Ακούγοντας τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, καμιά φορά αισθάνομαι σαν να βλέπω ταινία του Σέρτζιο Λεόνε. Για κάποιους από εμά, ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Και για κάποιους άλλους είναι για μια χούφτα δολάρια ο τίτλος της ταινίας που βλέπουμε. Από μια πλευρά λοιπόν θεωρώ ότι όλοι αυτοί που μίλησαν σήμερα ακολουθούσαν το σωστό δρόμο, όχι πάντα, αλλά από κάποιες οπτικές γωνίες. Δεν διορθώσαμε τα πάντα. Δεν διορθώσαμε όλα όσα έπρεπε να διορθωθούν στη γη και νομίζω ότι ο Επίτροπος ο κ. Κανιέτε θα επιστέψει εκ νέου με το θέμα, ας πούμε σε τρία χρόνια, όχι μόνο λόγω της Ενεργειακής Ένωσης, αλλά επειδή η τεχνολογική πρόοδος που βλέπουμε στον πραγματικό κόσμο για την ώρα πηγαίνει πολύ γρήγορα και δεν βλέπουμε πού θα καταλήξει και ποιες δυνατότητες θα έχουμε μετά από δύο ή τρία χρόνια. Λέγοντας ότι θεωρώ ότι διορθώσαμε ένα πράγμα, τι εννοώ. Εννοώ ότι ο φίλος μου Φιέλνερ το είπε. Είπε στα Σμπίλα Σπέρδεγκλε. Είπε ότι έχουμε σταθερούς ε, κανόνες του παιχνιδιού στα Σουηδικά. Αυτό που κερδίσαμε ήταν να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σταθερούς κανόνες για τη βιομηχανία. Διότι αν δεν το έχουμε αυτό, όσο πιο γρήγορη είναι η τεχνολογική εξέλιξη, τόσο μεγαλύτερο είναι ο κίνδυνο να κινηθεί προ άλλη κατεύθυνση η βιομηχανία. Νομίζουμε ότι αυτό το διορθώσαμε. Λέγοντα ότι διορθώσαμε, ταυτόχρονα όταν έχουμε πολύ ταχεία πρόοδο, ε, τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα. Ε, Επίτροπε Κανιέτε, λοιπόν, έχετε κάθε λόγο να ανησυχείτε κάπως θα έχετε πολλή δουλειά να κάνετε και θα επιστρέψετε σε εμά και θα προσπαθήσετε να διορθώσετε κάποια από τα επόμενα προβλήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και είμαι σίγουρο ότι θα έχουμε προβλήματα. Ευχαριστώ όλους σας, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και πώς να το πω, η μάχη συνεχίζεται. Ευχαριστώ. Κύριε Σιγητάκη, και συγχαρητήρια. Στις 12.30 ε, θα γίνει η ψηφοφορία και εδώ κλείνει η ζήτηση για αυτό το θέμα. Το επόμενο σημείο της ημέρας τη διάταξης. Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση.